Ήταν μια άσκηση μόνο αυτή, εκένωση κτηρίου. Και έτσι μπορούμε και πάλι να ξαναβρεθούμε και να συνεχίσουμε. Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η πρώτη από τις δύο εκθέσεις ΡΑΠΚΑΙ... όσον αφορά την ε, ασυλία του κ. Πάσκη. Δεν θα υπάρξει catch the eye, αυτό αποφάσισαν οι πρόεδροι των πολιτικών ομάδων. Οπότε αρχίζει η συζήτηση και ο κύριο Ζαπκά είναι ο πρώτος. Εισηγητή, βέβαια είναι ο πρώτος που έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσθέσω μία φράση μόνο στη συζήτηση επί της ημερησίας διατάξεως για την ασυλία ντεμαγκίστρης. Δεν προβλέπεται συζήτηση σε αυτό παρά μόνο ψηφοφορία. Θέλω να σας πω ότι ο ντεμαγκίστρης γενικώ έχει πέντε διαδικασίες εκ των οποίων εξετάζουμε τη μία η οποία δεν είναι αμφιλεγόμενη και στις επόμενες θα ακούσουμε πρώτα την άποψη του κυρίου Ντεμαγκίστρης. Σωστά, σωστά λέτε. Ήρεμα, το εξηγούμε αυτό, καμία πολιτική ομάδα δεν ζήτησε συζήτηση σχετικά με την κοινοβουλευτική ασυλία του κύριου Ντεμαζίστρης. Οπότε, όπως είπε ο κύριος Ραπτκάη, θα υπάρξει απλώς ψηφοφορία. Όμως, στην περίπτωση του κύριου Σπάσκιτς, η ομάδα των φιλελεύθερων και δημοκρατών ζήτησε συζήτηση. Και γι' αυτό ακριβώς και γίνεται η συζήτηση. Στην περίπτωση Ντεματζίστρης δεν ζητήθηκε συζήτηση. Και έτσι, όπως σας είπα κυρίες και κύριοι, η περίπτωση Ντεματζίστρης θα ψηφιστεί ευθύ αρχή. Οπότε βάζω και πάλι το χρονόμετρο στην αρχή. Κύριε Ραπκάη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απλούστατα το ήθελα να το διευκρινίσω διότι υπήρξε ένα σχόλιο από έναν συνάδελφο προηγουμένω. Ήθελα να πω ότι ο κύριος Σουσπάσκης επί του προκειμένου δεν έχει ασυλία διότι ε, στις 7 ε, Σεπτεμβρίου 2010 είχε αρθεί η ασυλία του κυρίου Σουσπάσκη και αυτό παραμένει. Ο κύριος Σουσπάσκη τώρα βάσει νέων στοιχείων στοιχείων ζητά να αποκατασταθεί η ασυλία του. Θέλω όμως να σας πω περί τίνος πρόκειται. Ο κύριος Σουσπάσκης κατηγορείται από τις ποινικέ αρχές της ε, Λιθουανίας ότι έχει ε, ε, κινηθεί, έχει παραπτώματα τα οποία άπτονται του, της κομματικής, κομματικά όταν ήταν αρχηγός του, του κόμματός του στη χώρα του. Μετά έγινε Ευρωβουλευτής ε, και το 2009 ε, έγινε Ευρωβουλευτής εδώ οπότε και απεκαταστάθη η ασυλία η οποία είχε αρθεί όταν είχε επανέλθει στη χώρα του σαν αρχηγός του κόμματος εκεί. Έχουν υπάρξει δύο συζητήσεις ή στην Επιτροπή μας. Δεν ξέρω αν ε, είναι αθώος ή υπέτειος ο κύριος Ουσπάση και είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζω και δεν είναι ε, δικό μου καθήκον να το αποφασίσω ούτε δικό σας. Αυτό θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη στη χώρα του, στη Λιθουανία. Εμείς πρέπει να δούμε αν υπάρχουν δύο απόψεις οι οποίες ε, ε, σημαίνουν ότι θα διατηρηθεί η ασυλία την οποία έχει ε, σαν Ευρωβουλευτής και θα υπάρχει διαφορετική ε, μεταχείριση από ότι ενός απλού πολίτη της χώρας τους. Και είμαστε πεπισμένοι ότι αυτό δεν ισχύει, διότι καταρχήν με αυτή την διαδικασία δεν μπορεί να εκφράσει ελεύθερα την γνώμη του δεν τον εμποδίζουν να εκφράσει ελεύθερα τη γνώμη του για θέματα φορολογικής νομοθεσίας. Επίσης δεν διώκεται για την πολιτική του δραστηριότητα. Αυτό είναι ίσως αμφισβητούμενο, αλλά αφού απευθύναμε ερωτήματα στις αρχές της Λιθουανίας, νομίζω ότι έχει ξεκαθαριστεί και το θέμα αυτό και πρέπει να άρουμε την ασυλία. Ο κύριος Σουσπάσικ έχει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πρωτοβάθμια και έχει ζητήσει να αναβληθεί η απόφαση μέχρι ότου υπάρξει μία πρώτη απόφαση. Αλλά απερίφθη αυτό εις το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τώρα ο κύριος Φάσικ μας λένε ε, νέα στοιχεία, μας λέει ότι υπάρχουν νέα στοιχεία, ότι τα στοιχεία του ε, διέρευσαν στο Wikileaks και παρακαλεί ε, να ε, αποκατασταθεί η ασυλία του. Εγώ τον προσπάθησα να τον πείσω να μην προβεί προς αυτή την κατεύθυνση, πράγμα το οποίο δεν δέχθηκε και όταν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέχτασε τα νέα στοιχεία είπε ότι ίσως για την ίδια διαδικασία στη Λιθουανία τα στοιχεία αυτά είναι σημαντικά αλλά όχι για την άρση της ασυλίας του. Άρα τον ακούσαμε λεπτομερώς σε πολλές συνεδριάσεις, συζητήσαμε και φτάσαμε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Δεν αποφασίζουμε εδώ αν είναι αθώος ή φταίχτης αλλά εάν έχει πρόσβαση στην ασυλία και δεν ε, μπορούμε ούτε να αποφανθούμε για το τι γίνεται ε, στη Λιθουανία ούτε αν ε, υπάρχει εκεί πολιτική δίωξη. Άρα εμένουμε στη γνώμη μας ότι διατηρείται η άρση της ασυλίας, δεν την άρουμε τώρα, είχε αρθεί η ασυλία και απλούστατα διατηρείται η άρση αυτή και αυτό σας προτείνω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Εκ μέρου των πολιτικών ομάδων τώρα, εκ μέρου του ΕΛΚ πρώτα απ' όλα, το λόγο έχει ο κύριος Βιέσκα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, είμαι μέλο της Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων με ιδιαίτερη χαρά εδώ και πολλά χρόνια. Όλο αυτό το διάστημα έχουμε εξετάσει δεκάδες και δεκάδες αιτήσει για άρση ασυλίας. Θέλω εδώ να υπενθυμίσω στους συναδέρφους ότι όπως είπε και ο συνάδελφος Ραπτκάη και το υπογραμμίζω και εγώ αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι διαφορετικό από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ξεκάθαρους διαδικαστικούς κανόνες όταν πρόκειται για την ασυλία των Ευρωβουλευτών και οι κανόνες αυτοί λένε ότι μπορούμε να αρνηθούμε την άρση ασυλίας μόνον εφόσον η συγκεκριμένη περίπτωση έχει να κάνει με την εντολή του εκάστοτε Ευρωβουλευτή. Με κάθε σεβασμό λοιπόν προς τον κύριο Ουσπάσκιτς και το έργο του ως ε, Ευρωβουλευτής, υπό την ιδιότητα του Ευρωβουλευτού, πρέπει να ξέρετε ότι μέσα στην ομάδα του ΕΛΚ το συζητήσαμε εκτενώς και μπορεί να συμπαθούμε τον κύριο Ουσπάστικ. αυτό είναι ένα θέμα, από την άλλη μεριά όμως οι κανόνες είναι κάτι άλλο, ο νόμος είναι κάτι άλλο. Εφόσον λοιπόν η συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει καμία σχέση με το έργο του κυρίου Ουσπάσκιτς υπό την ιδιότητα του Ευρωβουλευτού, δεν βλέπουμε γιατί να αρνηθούμε την άρση ασυλίας. Εξάλλου, ο κύριος Ραπτκάη εξήγησε την υπόθεση, εξήγησε περί την πρόκειται. Και εγώ θυμάμαι ότι πριν από λίγο πάνω από ένα χρόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε με την άρση ασυλίας του κύριου Σπάσκιτς. Τώρα να συζητήσουμε τώρα κατά πόσο απόφαση αυτή ήταν σωστή όχι, εγώ λέω πως ήταν σωστή. Ο κύριος Βότσον, εκ μέρους των φιλελευθέρων τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο κύριος Σπάσκετς είναι ένα περίεργο φαινόμενο στην Λιθουανία, γιατί είναι ρωσόφωνο και πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας και πολιτικός. Από την επιτυχία του απειλούνται άλλα πολιτικά κόμματα. Οπότε για μένα η υπόθεση αυτή είναι μια δίωξη βασικά γιατί χρησιμοποιούν ένα αστικό αδίκημα για να τον οδηγήσουν τελικά σε μια ποινική διαδικασία. Λοιπόν, η περίπτωση για μένα από τη στιγμή που ήρθε το αίτημα για άρση ασυλίας ήταν ξεκάθαρο. Ε, σιγά σιγά ήρθαν και άλλα στοιχεία όμως. Όχι μόνο η περίπτωση του Wikileaks, το οποίο αναφέρθηκε και ο κύριος Ραπτκάη, αλλά και ο τέος ε, Προσπρασάσκη δέχτηκε ότι ψηλά ιστάμενοι ε, κατηγορούν τον κύριο Σπάσκιτς γιατί απειλούνται. Και ξανά τώρα το ξανακούσαμε ότι πριν από πέντε χρόνια οι υπηρεσίες ασφάλειας πίεσαν τον πρόεδρο να πιέσει με τη σειρά του το δικαστήριο σε βάρος του κυρίου Ουσπάσκιτς. Και τώρα στην Επιτροπή πέντε άτομα στήριξαν ε, τον κύριο Ουσπάσκιτς νομίζω ότι αποτελεί έναν στόχο μιας εκστρατεία πολιτικής σε βάρο του για να αναγκαστεί αυτός και το κόμμα του να εγκαταλείψουν την πολιτική. Γι' αυτό λοιπόν ζητάω από του συναδέρφους να μην δεχτούν την άρση ασυλίας αλλά να την επαναφέρουν. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο ευχαριστούμε. Ο κύριος Τομασέσκη είναι ο επόμενος ε, ομιλητή εκ μέρου των ε, συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το θέμα που εξετάζουμε είναι περίπλοκο. Από την άλλη μεριά όμως είναι και σαφές. Γιατί σαφώς ο κύριος ε, Ουσπάσκιτς είναι θύμα μιας σκηνοθεσίας μεταξύ των ε, πολιτικών κομμάτων. Ο εισηγητής αντικατοπτρίζει την άποψη της σημερινής κυβερνητικής πλειοψηφίας στη Λιθουανία. Όμως, είναι οι ίδιοι εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να βγάλουν τον κύριο Ουσπάσκιτς από την πολιτική ζωή. Και νομίζω ότι ακριβώς αυτό είναι που περιπλέκει τα πράγματα και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο η ψηφοφορία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή κατέληξε έτσι όπως κατέληξε. Το ΕΛΚ ψήφισε όπως ψήφισε για το κύριο Λανσπέργκης είναι και αυτός αναμειγμένος στην περίπτωση. Όμως, ξεκάθαρα, δεν μπορεί να υπερισχύει ο πολιτσοφικισμός εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ πρόκειται για μια πολιτική υπόθεση και η ομάδα μου θα υπερψηφίσει, υπερ, θα ψηφίσει δηλαδή την ασυλία του κύριου Σπάσκη. Παρακαλώ κύριε και σαν εισηγητής βεβαίως θα ήθελα να λάβω το λόγο και έχω ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Δεν ήταν χαρά για μένα και πρέπει να σας πω τώρα ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι έκανε λάθος η πλειοψηφία και στην πρώτη και στη δεύτερη εξέταση στην πολιτική. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι ο πολιτικός ρόλος του κυρίου Σπάση στη πολιτική ζωή της χώρας του. Το θέμα είναι αν δικαιούται ε, να υπάρχει μία δίκαια διαδικασία ε, και αυτά που λέει ο κύριος Τομασεύσκη με το, ε, για τους Μολσεβίκους είναι κάτι το οποίο πρέπει να αγνοήσουμε. Εδώ δεν μπορούμε να πούμε αν ευθύνεται ή όχι. Το ερώτημα είναι έχει περιοριστεί ε, για τα, ε, τις πολιτικές του πεπιθήσεις ε, και το διώκεται λόγω των πολιτικών του πεπιθήσεων και στις δύο περιπτώσεις η απάντηση ήταν αρνητική και σας ζητώ να υπερψηφίσετε την έκθεσή μου. Ευχαριστούμε και τώρα κλείνει η συζήτηση και αύριο στις 12 θα ψηφίσουμε για τις εκθέσεις. Το επόμενο σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας, δηλαδή η προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2011. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συζητηθούν όλες οι διαφορετικές